Λίλους μια καλή επιστροφή. Α, ο κύριος Όντι για διαδικαστικό θέμα προηγουμένως. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι διαδικαστικό, είναι θέμα εφαρμογής των συνθήκων. Το έχω κάνει πολλές φορές τελευταίως. Ολοκληρώνεται η σύνοδος αυτή της Ολομέρειας. Σε 15 μέρες, πριν από 15 μέρες είχε γίνει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ήρθε, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Ε, και νομίζω ότι δεν είναι καλό ε, ένα όργανο σαν το δικό μας ε, που μπορεί να νομοθετεί να μην σέβεται την νομοθεσία αυτή. Προτείνω για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει 18 και 19 Δεκεμβρίου που θα έχει ε, την Ευρωπαϊκή άμυνα ως θέμα, το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές αυτό μέσω εκθέσεων που άλλωστε και σήμερα ψηφίσαμε, να καλέσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί μετά το Κοινοβούλιο και συνεπώς δεν θα μπορέσει να ε, έρθει να μας πει τι έγινε στο Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει να πω ότι βρίσκω θλιβερό να μην, να μην γίνονται σεβαστές οι συνθήκες Επίσης, νομίζω ότι δεν έχουμε αρκετές ανταλλαγές απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. ούτε ή άλλως, ούτε καν από τα, με τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούμε να έχουμε παρκείς ανταλλαγές απόψεων. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Οντή. Θα παραπέμψω στον αρμόδιο φορέα το θέμα αυτό στη συνέλευση των Προέδρων και θα σας ενημερώσω σε σχέση με τις αποφάσεις του σώματος αυτού. Και πάλι λοιπόν σας εύχομαι καλή επιστροφή.